Meine Damen und Κυρίες και κύριοι. Guten Morgen. Καλή σας μέρα. Ich bitte nicht so laut zu sprechen. Παρακαλώ μην μιλάτε τόσο δυνατά πρωί-πρωί. Για να μπορώ ήσυχα να συνεχίσω τον ύπνο μου. Λοιπόν, ερχόμαστε στο σημείο 13 της ημέρας της διάταξης. Κύριε Ντονζόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια έκθεση που έπρεπε να ψηφίσουμε σήμερα του κυρίου Ίντρικ Ταράντα σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και τον ρόλο της σε περιπτώσεις κρίσεων που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές και τις φυσικές καταστροφές και η οποία αφορά τη δικιά μας υποεπιτροπή. Φαίνεται ότι από αυτής τη εκθέσεως ε, πρέπει να γίνουν ακόμα περαιτέρω διαπραγματεύσεις για ορισμένες τροπολογίες. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω αναβολή της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Well, actually... It's true Αληθεύει αυτό που, που είπε ο κύριος Ντανζάν. Ε, ε, καθυστερήσαμε, δεν είχαμε καιρό στα έγγραφα γιατί τράβηξαν πολλοί διαπραγματεύσεις. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ε, είμαι υπέρ του να ε, μένουμε στο πρόγραμμά μας γιατί δεν είμαστε και δεν είναι και πολύ τα, ε, δεν είναι όπως τα ήθελα εγώ πάντοτε. Αλλά με αυτήν την αναβολή, σε συγκεκριμένη περίπτωση, πιστεύω ότι το ΕΛΚ θα έχει την ευκαιρία να προσεγγίσει την αρχική διατεωρχικό κείμενο και να αλλάξει γνώμη. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω τι θα κάνει το ΕΛΚ ως πρόεδρος της Επιτροπής, αλίμονο. Αλλά Βλέπω ότι επικρατεί συνένεση, οπότε και αναβάλουμε αυτό το σημείο της μέρας της δένταξης. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Και ερχόμαστε στην έκθεση της κυρίας Γιαννάκου. Για τα λεφτά, λέει ο πρόεδρος. Είναι εδώ, κυρία Γιαννάκου. Ποιος την εκπροσωπεί. Ποιο ε, εκπροσωπεί την κυρία Γιαννάκου για την έκθεσή τη. Hm? Έρχεται με μικρή καθυστέρηση η κυρία Γιαννάκου. Αν συμφωνείτε να ψηφίσουμε την έκθεση κυρίας Μπραντνερ πρώτη. Συμφωνείτε. Κυρία Μπραντνερ, παρατήρηση. Όχι, ευχαριστώ.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 αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 22 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έρχομαι στην 7 υπέρ, Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί τις τροπολογίες της εισηγήτριας μαζί με το συμβιβασμό. Από την 7 δηλαδή μέχρι τη 10 συν την κομπ. Είπε Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. Καταπίπτει. 13 είπε Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του έργου τέχνης. Äh, ja, Εγκρίνεται η έκθεση 57 ψήφι υπέρ 2 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια θερμά κυρία Μπραντνερ. Zurück. Επιστρέφουμε τώρα στο σημείο 13 της ημερησίας διάταξης. Ήρθε η κυρία Γιαννάκου και μπορούμε να αρχίσουμε. Κυρία Γιαννάκου, θέλετε να πείτε τίποτα πριν την ψηφοφορία. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι στην ε, τροπολογία 4 έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση ως εισηγήτρια και ότι υπάρχουν τέσσερις τροπολογίες ε, συμβιβασμού και δύο προφορικές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λοιπόν, γρήγορα με τις συμβαστικές τότε. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία συμβασμού 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 7 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. Η συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. Τώρα η 11 ψήφι υπέρ. Κατά απόχέ, απορρίπτεται. Τώρα 10 υπέρ. Κατά. Απόχες. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά στο ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη 12. Πέρασε. 16 υπέρ, 46 κατά. Εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρο. Αχ, συγγνώμη, απορρίφθηκε. Ερχόμαστε 13 επέ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 14 επέ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 με προφορική τροπολογία επέ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, το σύνολο της έκθεσης θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Λήξεις. Εγκρίνεται η έκθεση με ψήφους 59 υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια θερμά. Έτσι φαντάζεται κανείς την προεργασία από τον εισηγητή στις εκθέσεις. Ερχόμαστε στο σημείο 16 τώρα. Της κυρίας Κριστίνα Γιούλαντ για την υπόθεση Μαγνίτσκι. Σύσταση προς το Συμβούλιο. Η κυρία ο Γιούλαντ θέλει να πει τίποτα. Πριν περάσουμε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 Ε, για όσους ήταν εδώ στη χθεσινή συζήτηση για τις τροπολογίες θα καταλάβουν ότι υπάρχει ένα μόνο πρόβλημα με την έκθεση τροπολογία 10 συγκεκριμένα και διατύπωση που προτείνω εγώ στη δική μου τροπολογία. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Όγιλαντ καθώς και τον σίγουρα από πλευρά των σοσιαλιστών μπορούμε πλέον να συμφωνήσουμε με τις τροπολογίες και σας προτείνω με μια προφορική τροπολογία Λέει τώρα η παράγραφο. Ε, Θα ρίνει το Συμβούλιο να τηρήσει μια συνεκτική και προορατική στάση σχετικά με άλλε σοβαρέ παραβίασει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία με βάση καλά τεκμηριωμένων, σύγκλινουσών και ανεξάρτητων πηγών και πιστικών τεκμηρίων και να θεσπίσει παρεμφέρει περιοριστικά μέτρα κατά παραβατών ως έσχατο μέτρο τελεία. Das ist nicht der Fall, dann werden wir jetzt über den Antrag. Ε, ε, θα ψηφίσουμε αυτή τη ε, διατύπωση υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Η 11 σε δύο τμήματα, υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της σύστασης αρχίζει τώρα. Abstimmung ist geschlossen. 62 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κυρία Ογιουλάντ. Και τώρα Έχαμε στο σημείο 17. Συμφωνία εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου. Μία τροπολογία υπάρχει της κυρίας Λούνατσεκ υπέρ της απολογίας παριθμών 1. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο της γραμμοδότησης θα ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά. αποχές. Εγκρίνεται με 54 ψήφους υπέρ 9 ε, κατά και μία εποχή. Συγχαρητήρια κύριε Σαλαφράγκα. So, wir kommen nun zu dem Thema 18. τώρα στο σημείο 18 μια στρατηγική ψηφιακή ελευθερία στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Σάκε. Ποιο ζήτησε το λόγο, κύριο Σίβιτς. Πρόεδρε, πριν αρχίσουμε και ακούσουμε την παρουσίαση, θα ήθελα να δηλώσω έκπληκτος. Δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον, την εισηγήτριά μας αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να εκφράσουμε από πλευρά πολιτικών ομάδων τη θέση μας. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά αν μία μέρα ανακαλύψουμε ότι ε, σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε ένας πρέσβης ε, λόγω μια ταινία στο διαδίκτυο, τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι είναι σημαντικό το διαδίκτυο. Παρακαλώ να προβλεφθεί χρόνο για να συζητήσουμε τι εστί διαδίκτυο και τι είδους ευκαιρίες και κινδύνους όμω συνεπάγεται για την εξωτερική μα πολιτική πολιτική. Δεν ψηφίσαμε την έκθεση Τάραντ, αγαπητοί συνάδελφοι, γι' αυτό έχουμε περισσότερο χρόνο. Οπότε μπορούμε να συζητήσουμε ε, το θέμα εκτενέστερα από όσο έχει προβλεφθεί. Συμφωνείτε. Κερδίσαμε χρόνο γιατί δεν ψηφίσαμε την έκθεση Τάραντ που ήταν πολύ μεγάλη. Έχουμε λοιπόν κερδίσει περίπου μισή ώρα. Άρα μπορούμε να την αξιοποιήσουμε αυτή για τη συζήτηση. Κυρία Σάκε, παρακαλώ να είστε ε, σύντομοι για να έχει αρκετό χρόνο ο κύριος Σίβιτς. Μεγάλη μου χαρά, πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το πρώτο σχέδιο αυτής της έκθεσης ε, ε, για τις, για τις ελευθερίες στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια έκθεση που ασχολείται ειδικότερα για θέματα ασφάλειας και άμυνας στον κυβερνοχώρο ενώ αυτή τη στιγμή συντάσσεται και εξετάζεται στην Επιτροπή ΣΕΝΤΑ. Πρόεδρε, θα μπορούσατε να σβήσετε το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο θα δείτε ότι στη δική μου έκθεση αποδίδω έμφαση σε όλες τις υπόλοιπες ε, διαστάσεις εξωτερικής πολιτικής, εμπόριο, ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη, αναπτυξιακή πολιτική, διεύρυνση και ούτω καθεξής. Αυτό το πρώτο σχέδιο που έχετε στους φακέλους σας είναι το προϊόν συνεργατικής προσπάθειας ε, με άλλους σκιώδεις εισηγητές. Θέλω να τους ευχαριστήσω παρεπιπτόντως. Είναι όμως και το ε, προϊόν των διαβουλεύσεων από με την κοινωνία των πολιτών, ε, ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων που καλούνται να αντεπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα επιτόπου σε χώρες από την Κίνα μέχρι την Ινδία, από την Τινησία μέχρι το Μπαχρέιν, τη Λευκορωσία κτλ. Ο στόχο ε, της στρατηγικής είναι να εξετάσει και τις ευκαιρίε, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση, ε, για να αντιμετωπίσουμε ε, το, και να χειριστούμε το νέο ρόλο των νέων τεχνολογιών στη ζωή των ανθρώπων ανά τον κόσμο και πώς θα απαντήσουμε μέσω της πολιτικής μας. Ο στόχος λοιπόν της έκθεσης είναι να εκδώσουμε συγκεκριμένες συστάσεις για την κατάρτιση μιας πολιτικής για το ρόλο των νέων τεχνολογιών πληροφορικής ούτως ώστε να ενταχθούν ε, οργανικά μέσα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν στους ανθρώπους ανά τον κόσμο με μεγαλύτερη ελευθερία να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, να εκφράζονται ελεύθερα, άλλαξε η ελευθεροτυπία και είμαστε μάρτυρες πλέον διαφόρων παρεμβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί πλέον μπορούν να τεκμηριώνονται και να ε, είναι διαθέσιμε επιγραμμικά. Όχι μόνο σε σχέση βεβαίω με τα ανθρωπίνα δικαιώματα, ε, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των νέων τεχνολογιών, αλλά και σε σχέση με τι οικονομικέ εξελίξει, που είναι εξίσου σημαντικό αφετέρου. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερο οι τεχνολογίε ε, για την καταστολή και για να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα σε τρίτε χώρε. Βλέπουμε ε, όλο και περισσότερα ε, πρακτικές μαζικής ε, παρακολούθησης, ε, υποκλοπής, ε, τηλεφωνημάτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε και να παραδεχόμαστε τη σημασία των νέων τεχνολογιών και της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας έτσι ότι θα χρησιμοποιηθεί αυτή η νέα δύναμη για το καλό, δηλαδή για οικονομική ανάπτυξη, πολιτιστική ανάπτυξη και να μην συνιστά η νέα τεχνολογία απειλή για τους ε, ανθρώπους στην καθημερινή του ζωή. Έχω διάφορα κεφάλαια στην έκθεσή μου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το εμπόριο για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις σε σχέση με το ε, τι πρέπει να κάνουμε ούτω ώστε να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία. Παραδείγματο χάρη στον τομέα του εμπορίου εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνολογίε που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ χώρε όπου δεν υπάρχει κράτο δικαίου, όπου γνωρίζουμε ή μπορούμε να μάθουμε ότι ε, θα χρησιμοποιηθούν αυτέ οι τεχνολογίε για να ε, φημώσουν την ελευθερία τη έκφραση ε, για να παρεμβιάσουν ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε μεγαλύτερη λογοδοσία λοιπόν και διαφάνεια από πλευρά επιχειρήσεων επιχειρηματικής κοινότητας, καλύτερη συνεργασία με αυτήν ε, και κάνουμε συστάσει ε, στο πλαίσιο τη ε, Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη για αυτό το λόγο κτλ. Είναι επίσης σημαντικό στα πλαίσια των εμπορικών μας ε, συμφωνιών όπου είναι διαρκώς ε, ε, διωγούμενος ο ρόλος των νέων τεχνολογιών για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Οργανικός πώς έχει εξελιχθεί πλέον σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο όμως δεν έχουμε τόσους πολλούς κανόνες ή ρυθμιστικές διατάξεις που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία. Πώς να διακυβερνήσουμε το διαδίκτυο δηλαδή με την συμμετοχή των κοινωνίας των πολιτών των χρηστών των καταναλωτών που πρέπει να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις ούτως ώστε να είναι δημόσιος χώρος αλλά και εμπορικός χώρος στο διαδίκτυο ταυτόχρονα. Επίσης υπάρχουν διάφορες διεθνείς πλατφόρμες ε, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, όπως παραδείγματο χάρη η Διεθνής Τηλεπικοινωνιακή Ένωση και το Διεθνές Διαδικτυακό Φόρουμ, όπου αποστέλει αντιπροσωπείε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα το συνεχίσουμε διότι είναι μεγάλες οι προκλήσεις που εξετάζουν ε, τέτοιου είδους ε, ομάδε. υπάρχει μια απόπειρα για μαζική λογοκρισία, μαζική παρακολούθηση και χρησιμοποιείται από οικονομικής και πολιτικής ε, πλευράς πλέον η μόχλευση που έχουμε για να σταματήσουν αυτές οι κακές πρακτικές και ε, έχουμε εκδώσει σχετικές συστάσεις. Εφόσον έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε το θέμα, θα σταματήσω εδώ, αλλά κλείνοντας ε, θα έλεγα πως ε, πιστεύω ότι όλοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε και ευθύνη αλλά και ευκαιρία αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουμε ε, τη νέα στρατηγική για τις ε, ψηφιακές ελευθερίες στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προϋποθέτει ότι θα επιζητήσουμε αυξημένες γνώσεις και συνειδητοποίηση του ρόλου του διαδικτύου εφ' και Καλό θα ήταν να έχουμε πρόσβαση και στην πραγματογνωμοσύνη στο χώρο του διαδικτύου ε, για να επεξεργαστούμε τις τροπολογίες μας. Ε, με τα χαρά σε να δεχτώ οποιαδήποτε σχόλια έχετε, αλλά πάντως θα ήθελα να συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής με τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και με τους σκιώδεις εισηγητές, ούτως ώστε αυτή, αυτή η σημαντική διάσταση της εξωτερικής μας ε, πολιτικής και ιδίως στην αρμόδιοι επίτροποι για τα εμπορικά ζητήματα και για τα ζητήματα διαδικτύου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν των εργασιών μας ε, για να ρυθμίσουν ε, τις προκλήσεις ε, στους οικείους τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σίβιτς, πρώτος όντως. Σίβιτς. Dziękuję bardzo. Chcę wyrazić najpierw podziw dla E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ε, αποτελεσματικότητα με την αντιδράσατε ε, όσον αφορά την συζήτηση που ζήτησα επί του θέματος αυτού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την ε, άμεση αντίδραση αυτή. Να πω τα εξής λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ότι το διαδίκτυο είναι πλέον αναπόσπαστο τμήμα της ζωής μας. Δεν είναι πλέον επιλογή, δεν είναι κάτι περίεργο, κάτι ξένο, κάτι ιδιαίτερο η πολιτική πραγματικότητα, ε, αλλά και όλα τα άλλα στοιχεία της καθημερινής ζωής των ανθρώπων πλέον περνούν μέσα από το διαδίκτυο. Είναι κάτι που συμβαίνει είτε το θέλουμε είτε όχι. Είδαμε ας πούμε ότι στην Αραβική Άνοιξη ε, ξεσηκώθηκε ο κόσμος ε, μέσα από μηνύματα που περνούσαν από τα δίκτυα έτσι, κοινωνικής δικτύωσης, ε, από τα μέσα συγγνώμη, κοινωνικής δικτύωσης και επομένως πραγματικά αυτά είναι. Έτσι έχει η πραγματικότητα από την άλλη πλευρά μπορούν στο διαδίκτυο να κυκλοφορήσουν φιλμάκια τα οποία όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και το θάνατο ανθρώπων. Επομένως ναι, ελευθερία, ε, αλλά πώς, πώς ε, μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτόν τον χώρο. Έγινε μια προσπάθεια μέσω της άκτα Ε, και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν και το είδαμε και από τις αντιδράσεις ε, που είχαμε για την άκτα ότι δεν μπορούμε το θέμα αυτό να το ρυθμίσουμε χωρίς ε, να να το ρυθμίσουμε χωρίς ταυτόχρονα να προκαλέσουμε προβλήματα να προκαλέσουμε προβλήματα στον, ε, στον κόσμο που θέλει την ελευθερία του, που θέλει να κατεβαίνει στους δρόμους, που θέλει να συνεννοείται για να κατεβεί στους δρόμους. Την είδαμε, επαναλαμβάνω, την ε, κατάσταση με την ε, άκτα και τις διαμαρτυρίες που είχαμε. δεν θέλουμε να ελέγξουμε την ελευθερία του ίντερνετ, αλλά καταλαβαίνετε πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί παρόλα αυτά. Εγώ καταλαβαίνω ότι η συγγήτρια έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, εκπώνησε μια εργασία η οποία είναι τροφή για σκέψη. Και ελπίζω ότι αυτή η εργασία δεν θα μείνει κενό γράμμα, ότι θα υπάρξει μια συνέχεια και ότι τελικά θα φτάσουμε στις σωστές αποφάσεις όσον αφορά τον περιορισμό ε, της ελευθερίας σε αυτόν τον τομέα. Θα σας πω κάποιες σκέψεις που κάναμε στην ομάδα μου. Ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα από τα κεφάλαια της έκθεσης και βεβαίως είναι λογικό. Εάν θέλουμε να ρυθμίσουμε ε, κάτι τόσο σημαντικό όσο το διαδίκτυο, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να, ε, ε, αν θέλουμε να εισάγουμε νέες τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουμε μια αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα έχουν αυτές οι τεχνολογίες στους ανθρώπους. Ε, γιατί αυτές οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν πάρα πολύ εύκολα ε, την υποκλοπή των ε, τηλεφωνικών μηνυμάτων, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, είναι πάρα πολύ εύκολη η παρακολούθηση πλέον, επομένως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στην παράγραφο 32, εκεί που γίνεται λόγος για το, τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα προγράμματα ε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν και στα προγράμματα γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ε, να μην αναφερθούμε γενικά σε όλα τα προγράμματα, να πούμε και συγκεκριμένα σημεία στα οποία θέλουμε να στοχεύσουμε. Μία άλλη παρατήρηση να κάνω τώρα. Ε, υπάρχει και σχετική τροπολογία από την πλευρά μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι χρήστες του διαδικτύου είναι είναι ε, ε, γειτονέ μας, είναι συνομιλητές μας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε διάλογο. Ε, γιατί ξέρετε το ίδιο έγινε και με, την, ε, με τα αυτοκίνητα. Στην αρχή λέγαμε ε, τι ωραία που μπορούμε να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο με το αυτοκίνητο. Μετά τα αυτοκίνητα έγιναν πολλά και έπρεπε να υπάρχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και έπρεπε να ρυθμιστούν τα όρια ταχύτητας κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Κύριε Γκόμες, κύριε Πρόεδρε, πριν από 15 χρόνια βοήθησα να μηχανογραφηθεί μια περιοχή της ε, ε χώρας, ε, μια χώρα που λέγεται Ανατολικό Τιμόρ, που είχε γνωρίσει σφαγές και στις ορεινές περιοχές πήγα εγώ και βάλα κομπιούτερ. Και σήμερα έχουμε διαδηλωσμένα εκατομμύριο πολίτες ε, κατά αυτών των ηλιθείων μέτρων που σκοτώνουν την οικονομία μας. Δεν αμφισβητώ καθόλου την ε, σημασία ε, του διαδικτύου. αλλά τέσσερις πολίτες οργάνωσαν αυτή τη διαδίωση του εκατομμυρίου. Ούτε συνδικάτα, ούτε οργανωμένα σωματεία, ούτε πολιτικά κόμματα, ούτε κανένας άλλος. Και χάρη στην ε, ε, κοινωνική δικτύωση ε, έχουμε αυτά τα φαινόμενα και χρειάζεται διακυβέρνηση. Ε, βεβαίως και το διαδίκτυο. Είναι το ίδιο με την οικονομία. Πώς να το πω. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα χρειάζεται διακυβέρνηση και καθοδήγηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τη διαφορά και να δείξει ηγετικό. Και η Μαρίκη Σχάκ εδώ τα λέει πολύ ωραία. Ας πούμε, αναφέρεται στη σημασία για ε, τις ε, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, ε, πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι εταιρείες και αναφέρει μια σειρά δράσεων που δεν μπορούν να αποσυνδεθούν για να αποτρέπονται και να προλαμβάνονται οι καταχρήσεις. Δεν είναι μόνο η τρομοκρατία, είναι η κακοποίηση των παιδιών, η παιδική πορνογραφία, η κακοποίηση και των ηλικιωμένων. Τώρα πρόσφατα σκοτώθηκε ένας διπλωμάτης. Οι διπλωμάτες χάνουν τη ζωή τους για διάφορους λόγους, σε διάφορες στιγμές. Ε, ίσως γιατί ε, ε, υπάρχουν κάποιοι που υποκινούν τον όχλο κατά κάποιων άλλων ανθρώπων. Αλλά τώρα υπάρχει παγκοσμιοποίηση και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Τέλος, να πω ότι οποιαδήποτε στρατηγική και να έχει Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξωτερική της πολιτική, χρειάζεται οπωσδήποτε <coughs> να δρά εκ των προτέρων. Δηλαδή, όχι μόνο να υποστηρίζει ε, όσους είναι αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υφίστανται καταπίεση από αυταρχικά καθεστώτα, αλλά θα πρέπει ενεργά να τα πολεμά αυτά τα φαινόμενα και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και να την προωθεί για να μην φημώνεται η ελευθερία της έκφρασης όπως συμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και αυτό χρειάζεται η Ένωση, εκτός από τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε και την ανάγκη ε, σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλιώς η δική μας δημιουργή ε, πολιτιστικών έργων θα ε, μπλέξουν πάρα πολύ άσχημα. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> E, Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ε, ε, αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Σίβιτσε Πιο συγκεκριμένα όλες οι διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το σχέδιο ΑΚΤΑ μας ε, ευαισθητοποίησαν ε, για τα ζητήματα της ψηφιακής ελευθερίας. Από την άλλη πλευρά, ορθά είπε η συγγήτρια ότι οι νέες τεχνολογίες ε, έχουν πάρα πολύ σημαντική επιρροή από των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως από των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο διαδίκτυο, καθώς και για την ελευθερία των μέσων ε, μαζικής ενημέρωσης. Ακούσαμε πολλά απλά παραδείγματα ε, που το αποδεικνύουν στις συζητήσεις της Επιτροπής και στην Ολομέλεια. Τα παραδείγματα μας έδειξαν ότι στα κράτη όπου υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την διαδικασία εκδημοκρατισμού Ε, και παρότι υπήρξε απαγόρευση δημοσίευσης ε, κάποιων άρθρων, παρόλα αυτά κυκλοφόρησαν αυτά τα άρθρα ε, χάρη στο διαδίκτυο και έφτασαν στους αποδέκτες τους. Θα ήθελα να τονίσω ότι τον ιδιαίτερο ρόλο των κοινωνικών ΜΜΕ όπως το Facebook για την έναρξη της Αραβικής Άνοιξης. Όλοι όσοι ήθελαν ε, να φέρουν την αλλαγή στην Αίγυπτο οργανώθηκαν στο διαδίκτυο ε, και ο διοργανωτής ε, των εκδηλώσεων, των διαδηλώσεων, Αχμαρ Μασόφ, έλαβε και το βραβείο Ζαχάροφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικές είναι οι νέες τεχνολογίες για διάφορα κοινωνικά κινήματα. Αυτά που συνέβησαν στην Τινησία και στην πλατεία Ταχύρις στην ε, Αίγυπτο δεν θα ήταν εφικτά χωρίς ε, την, ε, τις νέες τεχνολογίες. Δημιουργείται ένα εικονικό δίκτυο ανθρώπων που υπεραμείνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιθυμούν την διάδοση ιδεών που έχουν ιδιαίτερη σημασία και ιδεολογιών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για αυτούς. Οι πάροχοι υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στο διαδίκτυο έχουν ε, τα δικά τους συμφέροντα. Γίνεται εκ μία συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη, πώς δηλαδή μπορεί να ενισχυθεί η αξιοπιστία ε, των επιχειρήσεων ε, για τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως ε, η χρήση του διαδικτύου. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνε στους επιχειρήσεις και πώς θα συνειδητοποιήσουμε και θα κατανοήσουμε όλες τις απειλές που ενέχονται στη διαδικασία. Όπως σωστά είπε η κυρία Γκόμες, οι απειλές σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία, με την οργανωμένη εγκληματικότητα που μεγενθύνεται χάρη στο διαδίκτυο. Πώς ε, λοιπόν να κατοχυρώσουμε την ελευθερία στο διαδίκτυο αφενός, ενώ ταυτόχρονα ε, θα ρυθμίσουμε τον τομέα για να μην υπάρχουν καταχρήσει και να περιορίσουμε δράσεις που είναι επιβλαβείς για το σύνολο της ε, κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να το συζητήσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Ιδιαίτερα δεδομένων των πιο πρόσφατων εξελίξεων. Και εγώ ε, δεν ξέρω πώς θα βρεθεί εδώ μια ισορροπία. Για μας η ελευθερία της έκφρασης είναι εκ των ουκάνευ, πολύ σημαντικό εργαλείο, για να μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και ο κόσμος ε, σε χώρες που κατά τα άλλα είναι αρκετά περιορισμένη η ελευθερία της έκφρασης. Είναι πολύ σημαντικό. αν επιτραπούν περιορισμοί για κάποιους λόγους, αυτό ε, μπορούν να το εκμεταλλευτούν κάποια καθεστώτα για να απαγορεύουν τελείω το διαδίκτυο. Ε, νομίζω ένα μεγάλο ε, πλεονέκτημα του διαδικτύου είναι ότι δρά διασυνοριακά και μπορεί να φτάνει μέχρι και σε καθεστώτα δικτατορικά. Από την άλλη, η ελευθερία της έκφρασης και του διαδικτύου βέβαια δεν επιτρέπεται να έχει τέτοιες συνέπειες. Μερικοί ανεγκέφαλοι να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να ε, δυναμητίζουν τον κόσμο. Δηλαδή ε, προκαλούν συνειδητά. Δεν είναι ε, ένα καλλιτεχνικό έργο που θέλουν να διαδώσουν. Απλούστατα θέλουν να υποδαβλήσουν τα μίση και τα πάθη μεταξύ θρησκειών και λαών. Εκεί είναι το θέμα. Πώς θα βρούμε ένα διεθνώς αποτελεσματικό ε, ένομο μέσο να κάνουμε τη διάκριση αυτών των δύο. Δεν έχω απάντηση σε αυτό, αλλά αυτό είναι το αποφασιστικό. Και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε μια νέα εφεύρεση και χρησιμοποιείται, έχει βέβαια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτό πώς μπορούμε να το φέρουμε σε μια λογική ισορροπία είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω αν στα πλαίσια της συζήτησης αυτής βρούμε καμιά ιδέα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει ε, να πάει με αστρονομική ταχύτητα αυτή η έκθεση, με την ησυχία μας να το συζητήσουμε. Με εμπειρογνώμονες, όχι τεχνικούς, αλλά εμπειρογνώμονες που να μπορούν ε, να συνδέσουν ε, τις αξίες, τη συνείδηση των αξιών με τη νομική υπόθεση. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερος χρόνος να το συζητήσουμε με την ησυχία μας, διότι όντως αυτό είναι σημαντικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, όπως είδαμε τώρα με την ταινία με το Μωάμεθ. Και με τα καλά της και με τα κακά της ε, αυτή η εξωτερική πολιτική και το εργαλείο δεν θα πρέπει να βιαστούμε με την ισχύ μας να το συζητήσουμε για να κάνουμε καλή δουλειά. Ε, το λόγο έχει η κυρία Σχάκε. Σας ευχαριστώ και εκτιμώ αυτά που είπατε για την ελευθερία την έκφρασης και για τη γενικότερη στάση μας ταυτόχρονα όμως θα, δεν θα πρέπει να τα πρόσφατα συμβάντα να επηρεάσουν καταλητικά τη συζήτηση. Θα ήθελα προς ενημέρωσή σας να αναφέρω ότι είχαμε ήδη στην ΑΦΕΤΕ τρία εργαστήρια για τα ανθρωπίνα δικαιώματα, το εμπόριο, τα ζήτηματα διπλωματίας, ε, τις ε, μεταγραφές ε, και μάλιστα πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είναι πολύτιμε πληροφορίε. Υπάρχουν μεταγραφές βιντεοσκοπήσεις Επίσης ε, μπορείτε να κρίνετε και από την εμπειρία σας ε, όσοι εργάζονται με τις νέες τεχνολογίες, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρενέβησαν σε αυτά τα εργαστήρια και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συζήτηση και να απαντήσω σε κάποια σημεία. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να διαπιστώσουμε ποιε είναι οι πλέον σημαντικέ στρατηγικές και με ποιο τρόπο μπορούμε να ενσωματώσουμε οργανικά σε όλες τις εξωτερικές δράσεις μας τις νέες τεχνολογίες. Με ποιο τρόπο είπατε εκπρόσωπο, στην υπηρεσία εξωτερική δράση μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποφύγει περιορισμό τους. Με ποιο τρόπο μπορούμε να ε, δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην στρατηγική non-disconnect που που έχουν καταρτήσει από κοινού η Επίτροπος Κρούς και η Πατή Εκπρόσωπος Άστον για τη χρήση των νέων τεχνολογιών Ε, επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο των ε, κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης όπως ε, το Facebook παραδείγματος χάρη είναι ένας χώρος συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων στο διαδίκτυο. Στην Αίγυπτο χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα για να βοηθήσει τους ακτιβιστές. Στη Συρία όμως πληροφορίες που ανταλλάσσονται σε ΜΜΕ κοινωνικά όπως το Facebook δυστυχώς παρεμποδίστηκαν από παρεμβατικές μεθόδους υποκλοπήσε και χρησιμοποιήθηκαν κατά των ακτιβιστών και των αντιφρονούντων. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, διαπιστώσουμε ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο και γενικότερες προοπτικές ε, για τον τομέα για να θέσουμε τους όρους όπου θα είναι ελεύθερο το διαδίκτυο, θα υπάρχει ελεύθερο εμπόριο στο διαδίκτυο χάρη στις νέες τεχνολογίες, επαναληφθεί το ζήτημα τη μαζική λογοκρισία, όπω στην Κίνα παραδείγματο χάρη, ζήτημα ιδιαίτερη βαρύτητα για μα, διότι δεν παρεμποδίζει μόνο την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά περιορίζει και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ω προ την αναπτυξιακή πολιτική, όπω είπε η κυρία Γκόμε, υπάρχουν ε, πολλαπλέ ευκαιρίε. Ε, για ε, πρόσβαση σε ε, σχετικά φθηνές ταμπλέτες και ηλεκτρονικά μέσα που τους εξασφαλίζουν πληροφόρηση και για ζητήματα που θεωρούνται ταμπού. Παραδείγματο χάρη τα δικαιώματα των γυναικών είναι δικαιώματα σεξουαλικής αναπαραγωγής με οι νέε τεχνολογίες έχουν επίση παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στι εκλογέ. Ε, για την παρακολούθηση των εκλογών και καταμέτρηση των ψήφων. Όμως, προσοχή, δεν πρέπει να ρυθμίσουμε υπερβολικά το διαδίκτυο μεγαλύτερες επιχειρήσεις ε, προτίθεται να συνεργαστούν μαζί μας για τη ρύθμιση του διαδίου, διαδικτύου, όμως προσοχή γιατί δεν χρειαζόμαστε πάντοτε απαραίτητα νέα νομοθεσία, νέους νόμους, ήδη έχουμε υπερβολικά πολλούς ε, σε ορισμένους τομείς, μπορούμε να εφαρμόσουμε τους νόμους που έχουμε στη διάθεσή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ανταγωνιστικότητα, για τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να τους εφαρμόσουμε τον τομέα των νέων τεχνολογιών. Θα πρέπει να κερδίσουμε ε, έδαφος στον τομέα αυτό. Θα συνεχίσω τις συζητήσεις με τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους βουλευτές που ενδιαφέρονται για το θέμα, αλλά και με τους χρήστες τους καταναλωτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς όπως οι επιχειρήσεις, ε, όπως ε, κάναμε μέχρι στιγμής ε, σε ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα στον κύβερνο κυβερνοχώρο. Νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Κελάμε στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ θα έπρεπε να καλύψει αυτά τα στοιχεία, ώστε να αποφύγουμε την επικάλυψη και να αλληλοσυμπληρώσουμε συμπληρώνονται οι εκθέσεις. Ωραία. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και κλεισμένο των θυρών. Θα παρακαλούσα όσοι σχολάτε τώρα να αποχωρήσετε. αφορά έτσι τις απίσω έδρανα αυτό που λέμε. Von hinten alle, die Berechtigung hier zu bleiben. Εκεί στα ορεινά δικαιούνται όλοι να παρευρίσκονται. Wir haben jetzt äh, die Diskussion mit Ακολουθεί η συζήτηση τώρα με τη νέα ε, πρέσβη στην Ιεμένη, την κυρία ε, Μούσαιτ. Ε, παρακαλώ, ελάτε εδώ στο Προεδρείο, κύριε Μούσαιτ.